έπρεπε να είναι ο κύριος Λούκα, αλλά δεν είναι εδώ. Ας περάσω στον επόμενο. Πώς πήσε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομο στην επεξήγηση ψήφου για την οικονομική ενίσχυση στην Ουκρανία την οποία θεωρώ ευπρόσδεκτη πέραν της πολιτικής υποστήριξης που προσφέρουμε μέσα από τις συζητήσεις μας στο Κοινοβούλιο διότι οθετήσαμε συγκεκριμένη μακροοικονομική βοήθεια 1,8 δις ευρώ με μέσο πρόθεσμο δάνειο. Πιστεύω ότι εάν θέλουμε να συνεχίσει το δρόμο της ε, δημοκρατίας του κράτους δικαίου, της μεταρρύθμισης αγοράς της Ουκρανία χρειάζεται να προσφέρουμε όχι μόνο πολιτική αλλά και οικονομική υποστήριξη για να μπορέσει να στηριχθεί όπως στηρίχθηκε η Ευρώπη από τις ΗΠΑ μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ελπίζω στο μέλλον να έχουμε να συστήσουμε άλλες μορφές ενίσχυσης. Και αυτό βέβαια θα πρέπει να ε, προχωρήσει παράλληλα με μεταρρυθμίσεις στην Ουκρανία ώστε να μην καταλήξουν τα χρήματα αυτά των ενισχύσεων στα, στις τσέπες ολιγαρχών αλλά να αξιοποιηθούν. Η κυρία Μορβάη για την ίδια έκθεση. Ευχαριστώ θερμά. Ο φίλος και συνάδελφος κύριος Μπάλτση δυσκολευθήκαμε να επιλέξουμε τη στάση μας στην ψηφοφορία για την έκθεση αυτή. Εμείς δε πολλό περισσότερο από ό,τι οι συνάδελφοι λυπή, επειδή είμαστε και Ούγγροι, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προσφερθεί βοήθεια στην Ουκρανική κυβέρνηση Ξέρουμε όμως ότι δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ε, ουγγρικής μειονότητας που ζει στην Δυτική Ουκρανία. Και γνωρίζουμε ότι είναι απάνθρωπες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι Ούγγροι οι οποίοι επιστρατεύονται, παρότι δεν τους αφορά αυτός ο πόλεμος, επιστρατεύονται στον Ουγγρικό στρατό. Ζουν σε συνθήκες φτώχειας, σαν να ήταν στον τρίτο κόσμο, με μισθούς Αφρικής με ένα ευρώ την ημέρα λίγο πολύ 30 ευρώ το μήνα συγκεκριμένα και κάτι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό Ακολουθεί ο κ. Μπάλζο Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ. Η Ουκρανία χρειάζεται την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, η μακροοικονομική οικονομική στήριξη, την οποία ψηφίσαμε και εγκρίναμε, δεν εξυπηρετεί τους ορθούς σκοπούς. Θα δαπανηθεί για να εφαρμοστεί το πρόγραμμα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ενώ εκεί υπάρχει πραγματική ανθρωπιστική κρίση και εκεί θα πρέπει να πάνε τα χρήματα που πάνε στην Ουκρανία. Όμως οι τροπολογίες μας απορρίφθηκαν από την πλειοψηφία της Ευρωβουλής. Πρέπει να σταθεροποιήσουμε την Ουκρανία. Γι' αυτό χρειαζόμαστε πρωτίστως την ειρήνη, ανακοχή, να πάψει η αιματοχυσία. Αυτά βέβαια είναι βραχυπρόθεσμες λύσεις για μακροπρόθεσμες λύσεις για την μακροπρόθεσμη εξασφάλιση της ειρήνης πρέπει να λάβουμε υπόψη τα συμφερόντα όλων των πλευρών. Ευχαριστώ. Μου φαίνεται ότι έχουμε γίνει πλέον Ουγγρικό Κοινοβούλιο εδώ, τμήμα του Ουγγρικού Κοινοβουλίου, γιατί οι, οι, οι μοναδικοί τρεις παρόντες βουλευτές είναι Ούγγροι. Ο κ. Ε, Μπόγκοβιτς ωστόσο είναι απόν. Το ίδιο και ο κύριος Μάμικινς. Ακόμα και το μικρόφωνο μου κλείνει, λέει η πρόεδρος. Τελευταία επεξήγησης ψήφου. Πάλι θα ήταν κανονικά ο κύριος Λούκα, αλλά είναι απόν. Η κυρία Μόρβαη λοιπόν. Πολύ δύσκολο μου φαίνεται να υπερψηφίζω τέτοια δημοσιονομικά μέτρα επιβολής φορολογίας. Νομίζω ότι Αυτά είναι ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Εμείς προσπαθούμε την έκθεση αυτή βέβαια να καταπολεμήσουμε την φοροδιαφυγή. Σύμφωνοι. Γνωρίζουμε και εκείνα τα θέματα των διαρροών του Λουξεμβούργου. Μιλούμε και για τον ίδιο τον κύριο Γιούνκερ εδώ, που ε, βεβαίω έχει εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ο οποίος κάνει ό,τι θέλει. Περί αυτού επρόκειτο. Δεν θα ήταν σωστό να βοηθήσουμε και άλλους. Για παράδειγμα, τα θύματα των ε, υποθηκών που λαμβάνονται σε άλλο νόμισμα και για τα οποία μίλησα πριν από λίγο. Και υπάρχουν βεβαίως και άλλες ε, συναλλαγές οι οποίες βλάπτουν τον απλό άνθρωπο και θα έπρεπε να είναι στο στόχαστρό μας. Ευχαριστώ αγαπητοί. Ο κ. Μπόγκοβιτς θα έπρεπε να λάβει το λόγο κανονικά αλλά είναι απόν τα πρακτικά της ε, συνεδριάσεως θα τα λάβετε στην αρχή της επομένης συνεδριάσεως δεν